Dear colleague, take your place. Please take your seat. We will start now. So we are... Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Η συνεδρίαση των συντονιστών είχε μια ημερήσια διάταξη πολύ βαριά και καθυστερήσαμε. Θα ανακτήσουμε τον χρόνο. Ζητώ συγγνώμη που καθυστερούμε, αλλά στις 5.30 θα πρέπει να συνεδριάσουμε από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, άρα πρέπει να είμαστε στην ώρα μας, έτσι ακριβής. Ξεκινάμε λοιπόν. Να σας πω καταρχήν ότι αποφασίσαμε τα εξή. Πρέπει καταρχάς να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη, αν δεν διαφωνείτε, εντάξει. Από εδώ και πέρα στις συζητήσεις μας θα έχουμε μία μέθοδο εργασίας που θα είναι η εξής. Αν δεν έχουμε αρκετό χρόνο, μετά τον εισηγητή μιλάνε ε, οι σκιώδεις εισηγητές. Και μόνο αν έχουμε χρόνο δίνουμε το λόγο και σε άλλους συναδέλφου. Έτσι, προχωρούμε τώρα. Έγκριση των πρακτικών, αν υπάρχουν παρατηρήσεις στα πρακτικά, να τι ακούσουμε, αλλιώ, προχωράμε. Όχι, εγκρίνονται τα πρακτικά. Έχουμε διερμηνία σε διάφορες γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά μπορείτε να μιλήσετε και να ακούσετε τα ελληνικά. Και βεβαίω ξέρετε πολύ καλά ότι μεταδίδεται στο ίντερνετ τη συνεδρίασή μα. Πάμε στο σημείο 5. Ο κύριος Γλέζος θέλει να μιλήσει. Ε, παρακαλώ, θα του δώσω το λόγο. Μια στιγμή, κύριε Γλέζο, μια στιγμή. Ένα λεπτάκι, έτσι όχι παραπάνω. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Προεδρείο, αγαπητή Πρόεδρε, έχω θίξει και το θέμα και άλλη φορά και ζητάω να γίνει ειδική συζήτηση από την Επιτροπή μας γύρω από το θέμα της ληστείας των αρχαιολογικών θησαυρών από το Τρίτο Ράιχ στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή το αίτημά μου είναι να οριστεί μέρα συζήτηση. Σήμερα, κύριε Κλέζο, θα πρέπει να μιλήσουμε για μια άλλη λαϊλασία που συμβαίνει στο Ιράκ και στη Συρία, έτσι. Θα κάνουμε και εκθέσει πρωτοβουλία για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε με του συντονιστέ αυτό το θέμα που προτείνετε εσεί και θα δούμε πώ θα καταφέρουμε να βρούμε μία ημερομηνία για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, έτσι. Δεσμεύομαι να το προτείνω στου συντονιστέ, θα ακούσω τι ε, απόψει του και θα δούμε. Θα δούμε ποιο θα είναι και το συγκεκριμένο θέμα πώς μπορούμε να το συζητήσουμε και πώς μπορούμε να παρέχουμε και ω κοινοβούλιο γι' αυτό. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο, στη συνάδελφο Διακόνου. Έχουμε την εξέταση του κειμένου για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Γίνεται μια γενική συζήτηση. Έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες μέχρι τις 30 Μαρτίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 16 Ιουνίου. Κυρία Διακόνου, έχετε το λόγο. Έχουμε 25 λεπτά το πολύ, 20 με 25 λεπτά για αυτό το θέμα, γιατί αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να τελειώσουμε στις 5.30. Ο κύριος Διακόνου, όχι η κυρία. Ε, Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης. Το έχουμε δημοσιεύσει εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Και για να κερδίσουμε χρόνο, θα παρουσιάσω μόνο τις βασικές ιδέες της έκθεσης. Εξετάζουμε δύο βασικά θέματα. Το ένα αφορά την πολιτική για την πολιτιστική κληρονομιά και το, το δεύτερο αφορά συγκεκριμένες λύσεις για τα ειδικά προβλήματα που εντοπίσαμε με τους εκπροσώπους ε, σε αυτόν τον κλάδο και τους ενδιαφερόμενους για αυτά τα θέματα. Η έκθεση ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το εξή. Καταρχάς, να εφαρμόσει την έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την πολιτιστική κληρονομιά και να εξασφαλίσει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ε, κλάδων και τομέων που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχουν διάφορες γενικές διευθύνσεις που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά, συμπληρώνουν τι δράσει η μία τη άλλη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεργάζονται καλύτερα, να συντονίζουν τι δραστηριότητέ του όταν εμπλέκονται θέματα πολιτιστική κληρονομιά. Χρειαζόμαστε λοιπόν συντονισμό σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων τη Κομισιόν. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή χρονιά αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά με συγκεκριμένο προπολογισμό. Εάν σχεδιαστεί καλά μια τέτοια πρωτοβουλία, μπορεί να προωθήσει την πολιτιστική κληρονομιά και μπορεί να δώσει πραγματικά εντυπωσιακού ε, καρπούς. Η Ευρωπαϊκή Χρονιά Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο προπολογισμό. και οι δραστηριότητες που θα οργανωθούν θα πρέπει να οργανωθούν και να υποβοηθηθούν από τα κράτη-μέλη. Επίσης, θα πρέπει οι πιθανοί δικαιούχοι να γνωρίζουν τι χρηματοδότηση υπάρχει για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω από διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές τις πληροφορίες είναι δημόσιες, αλλά υπάρχουν σε διάφορες ιστοσελίδες και παρουσιάζονται με πολύ τεχνοκρατικό τρόπο και μεταφράζονται σε κάποιες από τις επίσημες ε, γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι σε όλες. Είναι σημαντικό οι πιθανοί δικαιούχοι να έχουν μια πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Επίσης υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί και εμείς προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ζητάμε να δημιουργηθεί μία ενιαία δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα συλλέγει πληροφορίες για όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούν την πολιτιστική κληρονομιά και που θα διαιρεθούν σε τρεις βασικές βασικούς τομείς. Ε, δυνατότητες χρηματοδότησης, μια βάση δεδομένων παραδείγματα καλών πρακτικών και αριστείας στον τομέα, με τα link τα απαραίτητα, νέα και χρήσιμα links για τα προγράμματα και τις δραστηριότητες στον τομέα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την πολιτιστική κληρονομιά. Δεύτερον, θέλουμε να δώσουμε να κάνουμε ποιοτικά προγράμματα αποκατάστασης και ανακαίνησης και να έχουμε μηχανισμούς ελέγχου ούτως ώστε να αποτρέψουμε την ανεπίστρεφτη απώλεια της κληρονομιάς μας. Όλες αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να γίνονται με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, όπως αυτά που υπάρχουν στη σύμβαση της Γρανάδας και στο χάρτη της Βενετίας, ούτως ώστε να προστατεύσουμε την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Καλούμε την Κομισιόν να ξαναδεί το κατόφλι των 5 εκατομμύριων ευρώ για μικρής κλίμακας πολιτιστικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό κόστος αυτών των προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά μοντέλα διαφορετικής εναλλακτική ε, διαχείρισης και διακυβέρνησης, θα πρέπει να έχουμε νομικά ε, εργαλεία για εναλλακτική διαχείριση, ούτως ώστε να εμπλέξουμε καλύτερα τις τοπικές κοινότητες στις δραστηριότητε και προώθησης, αλλά και δια, διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς, το χάρη πρωτοβουλίες εταιρικών σχέσεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, όπου εμπλέκονται και τοπικές κυβερνήσεις. Δεν υπάρχουν όμως τα νομικά εργαλεία σε όλα τα κράτη-μέλη που επιτρέπουν τη δυνατότητα αυτή λειτουργίας αυτών των μοντέλων. Τώρα, το οικονομικό δυναμικό που έχει η πολιτιστική κληρονομιά. Η κληρονομιά μας έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει υψηλής ποιότητας βιώσιμες θέσεις απασχόλησης μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση τη ανεργία των νέων, εν μέρη. Και επίση τονίζουμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα τομέα που προσφέρει υψηλό δυναμικό θέσεων απασχόληση, μπορεί να είναι μια γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην, ε, και στην επαγγελματικό βίο, να δώσει μαθητείες ας πούμε σε νέους ε, και να τους απασχολήσει έτσι. Η πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο ρόλο στα επενδυτικά σχέδια του Juncker επίσης. Καλούμε τα κράτη-μέλη να ετοιμάσουν στρατηγικά προγράμματα για την πολιτιστική κληρονομιά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που θα είναι κατάλληλα. Θέλουμε να βελτιωθεί επίσης το μεθοδολογικό πλαίσιο, ούτω ώστε να έχουμε καλύτερες στατιστικές για την πολιτιστική κληρονομιά. Και στο τέλος η έκθεση τονίζει μία σειρά από ευκαιρίες που δεν θα πρέπει να χάσουμε. Συγκεκριμένα, προγράμματα κινητικότητας για ανθρώπους που δουλεύουν στον τομέα της πολιτιστική κληρονομιά. Θα πρέπει να προωθηθούν περισσότερο. Η ψηφιοποίηση τη πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίε στην έρευνα, θέσει απασχόληση και να προωθήσει και την οικονομική ανάπτυξη. Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συνεισφέρει επίση στην ανάπτυξη της ε, καλλιτεχνικής ε, δημιουργίας. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα όρια βέβαια εδώ των διαδικασιών που έχουμε. Περιμένω τώρα τις προτάσεις σας, τις τροπολογίες σας και η έκθεση θα ολοκληρωθεί μόνο όταν περάσουμε από όλα αυτά τα στάδια. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ελπίζω ότι συνεισέφερα σε αυτή τη συζήτηση. Ποιο ζητάει το λόγο από τους κοιόδης εισηγητές. Έχουν την προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ. Θα, θα σταθώ στα κύρια θέματα, όπως είπε η Πρόεδρος. Καταρχάς, θα ήθελα να σας συγχαρώ, κύριε εισηγητά, για την πλήρη έκθεση που μας παρουσιάζεται, που αντικειμενικά είναι μια σημαντική δουλειά που έγινε. Κάνετε μια σειρά από προτάσεις που έχουμε πει διάφοροι από εμά. Οι διάφορε έννοιες που αναπτύσσεται εδώ σίγουρα είναι αποδεκτές από τους σοσιαλιστές γιατί ο πολιτισμός είναι ένα κοινό αγαθό και έχει στρατηγικό δυναμικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά σημαίνει ότι προστατεύουμε την ιστορία μα, την ταυτότητά μα. αλλά και την ε, οντότητα του ευρωπαϊκού λαού που θέλουμε να φτιάξουμε. Πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πολύ σωστό είναι αυτό που είπε ο εισηγητή. Επομένω, η άποψή μα είναι γενικά θετική. Θα αναφέρω τώρα επιγραμματικά κάποια πράγματα. Συμφωνώ με το ότι θα πρέπει να έχουμε κατευθυντέ γραμμέ για νέες μορφές ε, συμμετοχική ε, διακυβέρνηση. Ε, να υπάρχει συνευθύνη στην κληρονομιά. Να υπάρχουν πιο έντονοι δεσμοί ανάμεσα στο τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και εταιρική σχέση μεταξύ δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ επίσης με την ιδέα να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό έτο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τονίσω γι' αυτό ότι είναι πολύ σημαντικό στην επόμενη διαδικασία του προπολογισμού, στον επόμενο προπολογισμό, το Κοινοβούλιο, εμείς ως συνομοθέτες, μαζί με το Συμβούλιο, να υποστηρίξουμε με πιστό την προσπάθεια της Κομισιόν και να έχουμε μια κατάλληλη χρηματοδότηση, όπως ακριβώς είπε ο εισηγητής. Άλλο σημαντικό είναι να υλοποιήσουμε αυτή την νέα ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την πολιτιστική κληρονομιά, που θα εμπεριέχει όλες αυτές τις πληροφορίες για τα προγράμματα χρηματοδότησης και που είπε ο εισηγητής. Και κάτι άλλο που θέλω να πω στον εισηγητή εδώ. Να αποφύγουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, ε, να λέμε ας πούμε να βουλιάξουμε πληροφορίες εκεί την ιστοσελίδα. Επίσης, υπάρχει, είναι σημαντική πηγή ιδεών η πολιτιστική κληρονομιά. Μπορεί να δημιουργήσει όμως και ε, υπηρεσίες, αγαθά, ε, δημιουργικές διαδικασίες που μπορεί να προστατεύσουν ε, και το περιβάλλον και τις αξίες του περιβάλλοντος. Επίσης θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ της επέκτασης του, πολιτιστικού τομέα και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, της φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Να πούμε πιο ρητά τη σχέση ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και την διάσταση της έρευνας και της καινοτομίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλών δεξιοτήτων. Και μία αμφιβολία στο σημείο 6 όπου μιλάμε για το ρόλο των κρατών μελών για να εξασφαλίσουν τον επαρκή έλεγχο της ποιότητας αλλά και της επαρκής επαγγελματικές δεξιότητες από αυτούς που κάνουν αναστήλωση των έργων τέχνης. Το θέμα είναι πώς θα εξασφαλίσουμε αυτή την ποιότητα. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε κάτι πιο σημαντικό, κάτι παραπάνω. Είναι σημαντικό επίσης να παρουσιαστεί μια τροπολογία για τη σημασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη δημιουργία ενός κανονιστικού γενικού πλαισίου για το επάγγελμα των ε, αναστηλωτών εργοτέχνης. Στηρίζω λοιπόν απόλυτα την, ε, την έκθεση αυτή και θα υποβάλω αυτές τις τροπολογίες μόνο έτσι συμπληρωματικά, για να τονίσω αυτά τα σημεία που σας ανέφερα. Πρόεδρος, θα δώσω το λόγο αποκλειστικά στους κοιότητες συζητητές λόγω χρόνου. Ζητώ συγγνώμη. Ή, εν πάση περιπτώσει, σε έναν ομιλητή, ένα ομάδα. Αλλιώς δεν έχουμε χρόνο. Κυρία Σουίντροβα, Eh, překladatelů a Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω ότι αυτή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Σνάρφο Διακόνου περιλαμβάνει πολύ σημαντικές τοποθετήσεις ό,τι αφορά την πολιτική κληρονομιά. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω αυτό το οποίο εγώ θεωρώ αναγκαίο και πρέπει να υπογραμμιστεί στην έκθεση. Θα κάνω και κάποιες συμπληρώσεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετική η πρόταση του συναδέλφου Διακόνου. Ιδίως ό,τι αφορά την άειλη κληρονομιά, επαγγέλματα, τον ζώντα πολιτισμό, αν θέλετε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως δεν δίνει έμφαση ακριβώς σε αυτό το σημείο στο ζωντανό πολιτισμό και ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι σημαντικός ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών για τους διαφόρους πολιτισμούς, όλα αυτά δεν αναφέρονται. Θα έχουμε και ακρόαση σχετική. Ο διαπολιτισμικός διάλογος λοιπόν είναι σημαντικός, είναι και ένα εργαλείο καταπολέμησης ε, του εξτρεμισμού και εντός Ευρώπης και εκτός Ευρώπης. Θα ήθελα επίσης ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σε τακτά διαστήματα έκθεση σε σχέση με την κατάσταση της ε, ηλικής και άλλης ευρωπαϊκής κληρονομιάς ε, με συστάσεις για το μέλλον. Ο εισηγητής παρουσιάζει ορισμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που χρήζουν βελτίωση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ε, πιστώσεις ε, ή τα δάνεια. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε και να μιλούμε για ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, θα πρέπει να είμαστε επίσης σε θέση να περιγράψουμε την κληρονομιά αυτή, να πούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και νομίζω ότι η περιγραφή ακριβώς της κατάστασης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ε, σε αυτό το στάδιο είναι κάτι το οποίο λείπει και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να αναλάβει αυτή την περιγραφή. Θα υποβάλω Σχετική τροπολογία λοιπόν και κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω είναι ότι είναι ανάγκη να έχουμε δείκτες Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να μας περιγράφουν την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς. Δεν έχουν καταρτιστεί τέτοιοι δείκτες όμως ε, μέχρι στιγμής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι λογικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στρέφεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Και σίγουρα θα διατυπώσουμε προτάσεις, ε, μέτρα και θα έχουμε και κάποια αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια άλλη μου πρόταση αφορά την ψηφιοποίηση. θα είπε και ο συγητής. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια πύλη όπου θα μπορούν εκεί να δημοσιεύονται πληροφορίες για το ενδεχόμενο χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σήμερα, σε επίπεδο UNESCO, υπάρχει το λεγόμενο Memory of the World, μνήμη του κόσμου. Είναι πολύ κατάλληλο εργαλείο αυτό. Καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει κάτι αντίστοιχο, το Memory of Europe, η μνήμη της Ευρώπης. Διότι έχει η Ευρώπη μια κληρονομιά πολύ σημαντική και θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να αναρτούν στοιχεία για αυτή την πολιτική κληρονομιά στη συγκεκριμένη πύλη. Και μπορεί αυτό να επηρεάσει θετικά και την αξία των ευρωπαϊκών μνημείων. Έχουμε και το ευρωπαϊκό σήμα ε, πολιτικής κληρονομιάς. Αυτά είναι λοιπόν τα αιτήματά μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να έχει και το ρόλο του συντονιστή κατά κύριο λόγο για να μπορούμε να μιλήσουμε για ευρωπαϊκή κληρονομιά. Ε, ευχαριστώ και ελπίζω να μην μακρηγόρησα πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Σφίτροβα. Ο επόμενος συνάδελφος. Ε, Ευχαριστώ, θα μιλήσω πολωνικά. Όταν ε, διάβασα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, πραγματικά σκέφτηκα πως πρέπει να ευχαριστήσω την... τον εισηγητή. Τώρα θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Θεωρώ πως θα πρέπει να γίνει κάποια αναφορά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί το πλαφόν πρέπει να ανέβει από τα 5 στα 10 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε και κάποιες αμφιβολίες για την πρότασή σας για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιστικής Κληρονομιάς. Έχουμε λοιπόν την εξής ερώτηση. Τι ε, ακριβώς θα είναι αυτό το έτος, τι θα γιορτάζουμε και ποια η διαφορά μεταξύ αυτής εκδήλωσης και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων. Ε, τώρα κάποια γενικότερα σχόλια μιλάτε για ψηφιοποίηση. Θα ήθελα να τονίσετε και τον ρόλο της παραδοσιακής ε, πρόσβασης. Είμαι πανεπιστημιακός, αντιλαμβάνομαι πως η ψηφιακή τεχνολογία και η πρόσβαση αυτή εκ του μακρόθεν δεν μπορεί πάντα να αντικαταστήσει τις ε, παραδοσιακές ε, μεθόδους. Αυτά τα οποία βλέπουμε στο ίντερνετ ε, δεν υποκαθιστούν την ζωντανή επαφή. Και υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο λείπει ο ρόλος ε, της ε, θρησκευτικής ε, κληρονομιάς στην Ευρώπη και πρέπει νομίζω να αναφέρετε και στην έκθεσή σας την ανάγκη της προστασίας της κληρονομιάς των μειονοτήτων, εθνικών, θρησκευτικών κτλ. Και επίσης των μεταναστών, οι Ευρωπαίοι μιλάνε πολύ για την κινητικότητα, ότι είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει νομίζω να συμπεριλαμβάνει και την δυνατότητα να προστατευτεί η πολιτική κληρονομιά των μειονοτήτων που ζουν ε, στην Ευρώπη και θα ήθελα επίσης ε, να σας πω, να αναφέρω μια διαφορετική ε, προσέγγιση. Μιλήσατε για την οικονομική σημασία της πολιτισμικής ε, κληρονομιάς. Ε, όμως ε, θεωρώ πως δεν θα πρέπει να βλέπουμε το πράγμα μόνο θεωρητικά. Πρέπει να αναφερθούμε στις μεθόδους χρήσης της κληρονομιάς. Δεν μπορεί δηλαδή να μιλάμε μόνο για τον τουρισμό. Παραδείγματο χάρη στην Πολωνία έχουμε την Κρακοβία. Η Κρακοβία έχει αναπτύξει τον τουρισμό, αλλά κάθε φορά που πάω αναρωτιέμαι σε ποιο βαθμό οι τουρίστες αυτοί εκμεταλλεύονται αυτέ τις ευκαιρίε που υπάρχουν για τον πολιτισμό. Ξοδεύουμε τόσα λεφτά καλό είναι να δίνουμε και κάτι για τον πολιτισμό, όχι μόνο για τις υποδομές. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μια καλύτερη υποπτία, γιατί που και που ανακύπτει ένα ζήτημα με την υποπτία, κάποια απάτη. Και τέλος. Κάτι για αυτή την ε, κεντρική προσέγγιση και τον συγκεντρωτισμό πρέπει να το αναφέρετε ε, νομίζω πως ε, που θεωρούμε ότι γίνεται καλύτερη διαχείριση του πολιτισμού στο κεντρικό επίπεδο ε, συχνά δεν ισχύει κάτι τέτοιο η Ευρώπη είναι πλούσια σε πολιτισμό και η προώθηση νομίζω αυτής της ε, κληρονομιάς ε, επαφίεται στους Ιταλούς, στους Πολωνούς ε, κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διευκολύνει αυτή την διαδικασία να μην έχει αυτές τις συγκεντρωτικές τάσεις. Καμιά φορά αυτοί που ζητάνε αυτή την κεντρική διαχείριση θεωρούν ότι μπορούν να ελέγξουν τον πολιτισμό δεν είναι τόσο εύκολο όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Κύριος Μαρεγκάλ έχει τον λόγο. καλησπέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντιακόν για την έκθεσή του. Είναι σαφή, συγκεκριμένη. Μα δίνει κάποιες μας δίνει κάποιες πολύ σαφές κατευθύνσεις και σε μεγάλο βαθμό συμμεριζόμαστε αυτές τις ε, τοποθετήσεις. Θα πρέπει βέβαια να προσθέσουμε δεχόμαστε και κάποια άλλα στοιχεία, πάντα βέβαια προσθέτοντας φιλοδοξία στο κείμενο. Συμφωνώ με τις απόψεις του τελευταίου συναδέλφου που έλαβε το λόγο και θέλω να πω ότι πέραν του να συνεχίσουμε και να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ε, πολιτική για την ενίσχυση των περιφερειών ε, και του ρόλου τους, που είναι και αρμόδιες περιφέρειες σε πολύ μεγάλο βαθμό για την ε, πολιτική κληρονομιά. Άλλωστε είναι ανεξάρτητες αυτόνομες. Είναι και ένα θέμα πόρων βέβαια, αλλά οι περιφέρειες και τα κράτη είναι αυτά τα οποία αναλαμβάνουν την πρόθεση πολιτικής. Αλλά η ίδια πολιτική κληρονομιά είναι μια ιδέα, είναι μια αρχή και θα πρέπει να δούμε αν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν κάποια στοιχεία άλλων και υλικών ε, μνημείων η πολιτική κληρονομιά. Χωρί να κάνουμε αλληλεπικαλύψει, υποκατάσταση ή να συγκεντρώσουμε το οτιδήποτε. Όχι. Σε κάποια περίπτωση απλά να δώσουμε δύναμη σε αυτό που μα ενώνει και να το προωθήσουμε. Επίση, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετεί στη δική της πολιτιστική πολιτική, ναι με να στηρίζει προγράμματα, εργαλεία ε, που στόχο έχουν ε, τη συμπλήρωση και τις ανταλλαγές, αλλά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε σε συγκεκριμένα κράτη, ιδίως κάποιες περιφέρειες, ε, να γίνουν θύμα του ίδιου του του πλούτου, της πολιτικής κληρονομιάς δηλαδή, γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν τόσο πυκνή, ποιοτική, πολυσύκληρονομιά κληρονομιά που με τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους πολύ δύσκολα μπορούν να τα καταφέρουν. Γι' αυτό χρειάζεται ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό ρόλο το ευρωπαϊκό επίπεδο. Να μιλάμε λοιπόν για ε, διπλασιασμό των πόρων, καλό είναι αυτό, αλλά να ορίσουμε και κοινούς στόχους. Από πέντε δις εγώ ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω επιγραμματικά να αναφέρουμε κάποια ζητήματα που θα μπορούσαν στο πλαίσιο της έξης να ληφθούν υπόψη ή να προσθεθούν στα αιτήματα της Ευρωπαϊκή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής σε θέματα πολιτικής κληρονομιάς. Θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα ε, το ευρωπαϊκό ε, καλό, ή κοινό συμφέρον. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι αυτά τα μνημεία ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και όπως υπόθηκε από μία συνάδελφο, ίσως και ένας κατάλογος δικτών θα ήταν χρήσιμος. Δεύτερον, να αναφέρω τρία ή τέσσερα στοιχεία για την άλλη κληρονομιά. Γρήγορα, γρήγορα. Κοινή ιστορία. Πρέπει να δουλέψουμε, να ερευνήσουμε, να απεικονίσουμε, να εφαρμόσουμε προγράμματα που έχουν να κάνουν την κοινή ιστορία των ευρωπαϊκών λαών. Ιστορικές διαδρομές, για παράδειγμα, που θα μας κάνουν να γνωρίσουμε και τις ε, λαμπρές αλλά και τις ε, σκοτεινές σελίδες της ιστορίας μας. Δεύτερον, γλώσσες. Πρέπει να επενδύσουμε στην προστασία ε, των γλωσσών και στην επικοινωνία μεταξύ αυτών, γιατί οι γλώσσες ε, είναι το χαρακτηριστικό της πολιτικής πολυμορφίας της Ευρώπης. Τρίτο, πάντα στο πλαίσιο τη άλλη κοινωνία πόλη, Η Ευρώπη ορίζεται μέσω της ε, προσφοράς και της συμβολής των πόλεων που την απαρτίζουν. Είναι ένα σύνολο, αλλά όχι απλό άθροισμα των πόλεων που την απαρτίζουν και κάτι παραπάνω. Τέλος, νομίζω ότι υπάρχει ένα στοιχείο που πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι και στην έκθεση και μπορούμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό, δηλαδή να έχουμε προγράμματα επιμόρφωσης των επαγγελματιών, ειδικά σε θέματα πολιτικής κληρονομιάς. Και ολοκληρώνω με μία σκέψη σε σχέση με αυτά που έλεγε ο κύριος Γλέζος, αλλά όχι μόνο. Η Ευρώπη έχει μία ευθύνη διότι έχει συγκεντρώσει και τεράστια πολιτική κληρονομιά προερχόμενη όμως από μη ευρωπαϊκές χώρες. Και πρέπει να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη ως Ευρώπη και είναι νομίζω και μια δυνατότητα που έχουμε να βελτιώσουμε ίσως και να ανασυγκροτήσουμε τις σχέσεις μας με άλλες χώρες. Ε, δεν μπορούμε να διαχειριζόμαστε μόνο το απεικιοκρατικό μας παρελθόν, αλλά να διαχειριζόμαστε και το παρόν μας. Τι σημαίνει ε, αυτή η πολιτική κληρονομιά για τις χώρες από τις οποίες προέρχεται. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κοινέ πολιτικές με τις χώρες αυτές και για τη διατήρηση της πολιτικής κληρονομιάς, ενίοτε και, και για την επιστροφή ορισμένων πολιτιστικών μνημείων στο φυσικό χώρο που ανήκουν. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Gracias. Ευχαριστούμε. Ο, η κυρία Ατινόλθη. Ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Θα είμαι λοιπόν λακωνικότατη. Σας ευχαριστώ την προσοχή σε δύο θέματα μόνο. Πρώτον, να μην θεωρήσουμε τα πολιτιστικά αγαθά ως ε, μέσο για να δημιουργήσουμε απλώ θέσεις απασχόληση. Το να θεωρήσουμε τα πολιτιστικά αγαθά και την πολιτιστική κληρονομιά ως, μια, ως ένα τουριστικό πόλο έλξης μπορεί να γίνει επικίνδυνο πραγματικά. Αντίθετα, θα πρέπει να τα θεωρήσουμε ως μέσο για να αναπτυχθεί ο πολίτης, ως πολίτης, να αναπτυχθεί η συνείδησή του. Και ενώ δίνουμε μεγάλη προσοχή στα σχολεία, όταν υπάρχουν ας πούμε φοιτητέ, οι πιο νέοι δίνουν σημασία σε αυτά τα θέματα στην πολιτική στην κληρονομιά όσο ε, μεγαλώνουν σε ηλικία αυτά τα άτομα και πηγαίνουν ας πούμε στο πανεπιστήμιο, ξεχνάνε λιγάκι, σαν αποσυνδέονται από τον πολιτισμό. Αυτή η κληρονομιά ε, δεν είναι μόνο για να δημιουργήσει ανάπτυξη ή εισόδημα. Θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε, να την κρατήσουμε, να την διαφυλάξουμε και για τις, νέ, για τις επόμενες γενιές. Επίσης, δεύτερο θέμα, έχουμε ένα πρόβλημα κονδυλίων, έτσι. Όποιος ξέρει, όποιος έχει επαφή με αρχαιολόγους, ε, με συντηρητέ έργων τέχνη, με φόρου μουσείων, ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν ε, χρήματα εκεί. Για τη διατήρηση των μουσείων, για τη διατήρηση των εργοτέχνη. Ε, υπάρχουν πολιτιστικά αγαθά, υπάρχουν εκκλησίε. Υπάρχουν πολιτιστικά, αρχαιολογικά αγαθά που είναι εγκαταλελειμμένα. Αν έχετε κάνει έτσι ταξιδάκια στην Ευρώπη, θα έχετε δει, α πούμε, εγκαταλελειμμένα αρχαιολογικά μνημεία. Τα οποία είναι θύματα βανδαλισμού, κλοπής, ακόμα, ακόμα. Εάν δεν υπάρχουν πόροι λοιπόν και αν δεν έχουμε νέου πόρου για την συντήρηση και την αξιοποίηση αυτών των μνημείων, θα παρακολουθούμε ανίσχυροι στην απώλεια αυτών των πολιτιστικών αγαθών. Αυτή είναι η μοίρα, η μοίρα μας. Σας ευχαριστούμε και για την λακωνικότητα. Η Κομισιόν είναι παρούσα. Κυρία, η κύριε Τζαμπιέρη, θέλετε να πείτε κάτι? Ο κύριο Τζαμπιέρη. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαιρόμαστε πολύ που μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη συνεδρίαση Βάλτερ Ζανπιέρη λέγομαι και είμαι στη υπεύθυνος για την ε, πολιτιστική πολιτική στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση του κυρίου Διακόνου είναι πολύ καλή, σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορούμε να την υποστηρίξουμε, θερμά μάλιστα. Σίγουρα καλό είναι να εργαζόμαστε διυπηρεσιακά και αυτό και κάνουμε άλλωστε Έχουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και πρέπει να σας πω ότι και οι συνάδελφοι από τη ΓΑΜΑ έχουν ε, συνεργαστεί και έχουν εκπονήσει μια έκθεση για την πολιτική κληρονομιά στην Ευρώπη που στόχο έχει να μας κατευθύνει για τους επόμενους διαγωνισμούς ε, και τα επόμενα προγράμματα στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020. Θα δώσω ε, κάποια στοιχεία και στα μέλη της Επιτροπής σας, στον εισηγητή, στην Πρόεδρο για να τα διαβάσετε, αλλά θα σας κάνω και κάποια ε, μικρή εισαγωγή. Ε, ακούσαμε την αναμόρφωση και ανάπλαση των αστικών χώρων, πολιτιστικό τοπίο. Αυτά είναι προτεραιότητες. Η χρηματοδότηση, η επιχειρηματικά μοντέλα, πιο κατάλληλα για την πολιτική κληρονομιά, είναι κάποιες από τις προτάσεις. Υπάρχουν πολλέ πρωτοβουλίε που αναλαμβάνουμε για να στηρίξουμε την πολιτιστική πληρωμιά. Πέρυσι δημοσιεύσαμε μια ανακοίνωση, η οποία συνοδευόταν και με τη χαρτογράφηση που στόχο έχουμε να επικαιροποιούμε και εκεί θα βλέπετε όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι θα ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι. Θα υπάρχει και πύλη ειδική, ένα πόρταλ από τη ΓΑΜΑ Βλέπουμε επίσης ε, ποια προγράμματα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Culture και από το πρόγραμμα Creative Europe, Δημιουργική Ευρώπη. Σίγουρα θα μπορέσετε να πάρετε πολλές πληροφορίε για πολλά έργα, πολλά project που υπάρχουν. Αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τα κράτη-μέλη, γιατί φυσικά είναι κοινή, μεικτή αρμοδιότητα, ε, το ακούσατε και από συναδέλφους σας ε, Δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη τα οποία πρέπει να φροντίζουν για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των πολιτικών τους ε, μνημείων. Έχουμε όμως και ένα είδος συμμετοχικής διακυβέρνησης ε, οργανώσει μαζί με τα κράτη-μέλη. Συλλέγουμε καλές πρακτικές ήδη από φέτος και του χρόνου θα δούμε και τα επαγγέλματα της πολιτικής κληρονομιάς για να δούμε πού είναι τα ισχυρά, ποια είναι τα τροτά σημεία, πού πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο, τι πρέπει να κάνουμε περισσότερο για συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Δύο ακόμη σημεία, πολύ σύντομα. Η συζήτηση για τα διαρθρωτικά ταμεία φενός είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται και έχει να κάνει με αυτό το κατόφλι των 5 δις. Ορίστηκε αυτό το κατόφλι γιατί υπάρχει και στον κανονισμό ο ε, μικρής κλίμακας ε, έργα πρέπει να χρηματοδοτούνται και στο ομάδα εργασίας για τα εδερφωτικά ταμεία όμως το συζητούμε το θέμα αυτό του προπολογισμού. Υπήρχε ανάγκη όπως είπα γιατί το πρόβλημα ο κανονισμός να οριστεί αυτό το κατόφλι, αυτό το όριο. Μας εξήγησαν πού έφτασαν, ε, πώς έφτασαν στο ποσό αυτό. Υπάρχει και ένας περιορισμένος βαθμός ευελιξίας υπό την έννοια ότι Υπάρχουν πολλές υποδομές μικρής κλίμακας που μπορούν να ενταχθούν σε ένα έργο ευρύτερης κλίμακας. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να επεκταθώ γιατί η συζήτηση συνεχίζεται με τα κράτη-μέλη και τους συναδέλφου μα από την Κομισιόν. Τέλος. Δυο λόγια για τον ποιοτικό έλεγχο. Φυσικά και στηρίζουμε ε, τα έργα, τα project να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα. Τουλάχιστον όμως σε επίπεδο διαρθρωτικών ταμείων υπάρχει μεικτή διαχείριση, δηλαδή τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια και πρέπει να φροντίσουν ότι υπάρχει ποιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρακολουθήσει, έχει ένα, ένα ρόλο, αλλά δεν είναι δική μας η ευθύνη, είναι ευθύνη των κρατών μελών. Την πρόσκληση πάντως του κ. Διακόνου την αποδεχόμαστε με τα χαράς. Προσπάθησα να καλύψω όλα τα σήμερα, δεν ξέρω αν μου ξέφυγε τίποτα. Αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ε, ε, είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση, ενδιέφερε πολύ τους συναδέλφους. Οι τροπολογίες θα πρέπει να παρουσιαστούν ε, μέχρι τις 30 Μαρτίου 12 η ώρα. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους ε, που γίνονται έτσι τα πράγματα, αλλά έχουμε 25 λεφτά για να κάνουμε τρει, ακόμα συζητήσει για τρία διαφορετικά θέματα. Δεν υπάρχει χρόνο. Αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή χρονιά θα πρέπει να μιλήσουμε για πολιτιστική κληρονομιά που περιλαμβάνει και το περιβάλλον και να υπάρχει και μια διεθνή συνεργασία και διεθνείς σχέσεις ε, για να προστατευτεί το πολιτιστικό, περιβλα... το πολιτιστικό περιβάλλον. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον είναι το θέμα των αρμοδιοτήτων. Έτσι. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ποιος έχει αρμοδιότητα γιατί σε αυτόν τον τομέα. Και εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη μεγάλη ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ε, πολιτιστικές διαδρομές. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για μια σύντομη απάντηση, αλλά δεδομένου του πολύ συχτού χρονοδιαγράμματος, ένα λεπτό, ένα λεπτάκι μόνο, έτσι. Μια και το λέτε στα Ιταλικά, ένα λεπτάκι μόνο σας δίνω. Πολιτιστική κληρονομιά σημαίνει επιστροφή των έργων τέχνης στον χώρο δημιουργίας τους. Δεύτερον, αναστήλωση των έργων τέχνης. Τρίτον, πολιτιστική λειτουργία που σημαίνει πέρα από την πόλη πρωτεύουσα και πρωτεύουσα περιοχής και πολιτιστικό χωριό. Η μέθοδος για αυτό το λόγο είναι τα κονδύλια προς αυτές τις κατευθύνσεις η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή την προσπάθεια όπως είπε ο συνάδελφος Μοργάνο και η πολιτιστική παιδεία και συνείδηση όπως είπε η Ισαβέλα Αντινόλφη. Ε, Ένα λεπτό. Μία κουβέντα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις συνεισφορές σας, για όλα τα σχόλιά σας. Περιμένω τις τροπολογίες σας. Και κάτι που μοιάζει σαν αστείο, αλλά είναι αλήθεια. Περιμένω τις τροπολογίες ε, για να τις ενσωματώσω στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση γνωμοδότησης Ernest Μαραγκάλ ενίσχυση τη θέση των κοριτσιών μέσω τη εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρμοδιότητα τη επιτροπή ΦΑΜ. Έχουμε μέχρι τι 30 Μαρτίου 12 η ώρα για τι τροπολογίε και θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον ίδιο τρόπο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομο, πιο σύντομο από ό,τι πριν θα είμαι. Πρόκειται για γνωμοδότηση στην προκειμένη περίπτωση από την ε, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας γνωμοδότηση σε έκθεση της Επιτροπής ε, Γυναικών. Όπως γνωρίζετε, αντικείμενο είναι η ισότητα των φίλων στην εκπαίδευση. Τον μηχανισμό χειραφέτησης ε, εν γέννη ή ενδυνάμωσης της γυναίκας και ιδίω ποιος είναι ο ρόλος εκπαίδευσης. Στη δική μας νομοδότηση ξέρετε ότι έχουμε κάποιους περιορισμούς Μπορεί να είναι μακροσκελέ στο κείμενο, φυσικά και μπορεί να κατατεθούν ε, τροπολογίε. Τέσσερι ιδέε λοιπόν περιλαμβάνει. Μία αναφορά που είναι και στην έκθεση τη κυρία Ροντίγκε, που είναι η καθήλυνα αρμόδια, την Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών. Αναφορά λοιπόν στα στερεότυπα των ε, φύλων που παραμένουν στα εκπαιδευτικά συστήματα. Η παρουσία αυτών των ε, στερεοτύπων είναι βέβαια κάτι αρνητικό, το οποίο το κατακρίνουμε και υπάρχει σε όλου του τομεί Μιλάμε και για τη διδακτέα ύλη ε, και το πρόγραμμα σπουδών, αλλά και γενικότερα ε, στο εκπαιδευτικό έργο. και επηρεάζει τις επιλογές κατάρτισης ε, και επαγγελματικού προσανατολισμού των γυναικών. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο θέμα, στερεότυπα εν γέννη. Δεύτερον, ποιος είναι ο ρόλος της άτυπης εκπαίδευσης και πώς αντικατοπτρίζεται στα εκπαιδευτικά συστήματα για πολλές γυναίκες, πολλά κορίτσια στην Ευρώπη και πόσο μάλλον εκτός Ευρώπης υπάρχει ένα πάρα δευτερογενές αποτέλεσμα ε, σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό επίπεδο. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τις επεπιθείς παραδοσιακές πρακτικές που μπορεί να επιβάλλουν περιορισμού στην εκπαίδευση για τα κορίτσια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά να τα ε, αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα πρέπει να σεβαστούμε τι διάφορε πεπιθήσει και παραδοσιακέ ε, πρακτικέ, αλλά θα πρέπει να εγγυηθούμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα κορίτσια. Και ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη επιβολές διάφορες λόγω θρησκείας, ε, φιλής ε, κτλ. Πρέπει και αυτό να το λέμε υπόψη, αν θέλουμε να έχουμε ισότητα στην εκπαίδευση. Τρίτον, εκπαιδευτική. Είναι και αυτή πολύ σημαντική για την ε, καταπολέμηση των στερεοτύπων. Πρέπει να προωθήσουμε την εκπαίδευση των δασκάλων και των καθηγητών και από αυτό θα βασιστεί σε πολύ μεγάλο και επιτυχία της πολιτικής μας ε, για την αλλαγή τη κατάσταση. Αν λοιπόν εγκριθούν και από τα κρατημέλια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια μέτρα, θα πρέπει αυτά τα μέτρα να εφαρμοστούν και για την επαγγελματική και για τη διαβίου μάθηση, την εκπαίδευση των ενηλίκων άνθρωποι, γυναίκες που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν σπουδέ του ή υποχρεώθηκαν να τι εγκαταλείψουν, να μπορούν να τι συνεχίσουν. Είναι άλλωστε αυτό σύνηθε φαινόμενο στις χώρες μας. Αυτά περίπου λέει η έκθεση γενικέ ε, γραμμέ, και σίγουρα θα εμπλουτιστεί με τις δικέ σα ε, τροπολογίες και θα έχουμε και επαφή με την εισηγήτρια από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, ε, ελπίζοντας ότι θα στείλουμε ένα πολύ καλό μήνυμα για τις γυναίκες σε αυτό το τομέα της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε τον κύριο Μαραγκάλ. Θα δώσουμε το λόγο στους κοιόδης ε, εισηγητές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εκπαίδευση, όπως είπε και ο εισηγητής, είναι ένα μέσο σημαντικό για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών. Να βελτιώσουμε την οικονομική τους και κοινωνική τους θέση και να ε, έχουμε και κοινωνικές δράσεις πιο υπέρ των γυναικών. Τα, τα στερεότυπα, η φτώχεια ε, επηρεάζουν άσχημα τα, τις εκπαιδευτικές επιπτώσεις και άρα και την ένταξη μετά στον χώρο απασχόλησης. Σίγουρα ε, σε τεχνολογικούς και επιστημονικούς τομείς ε, δραστηριοποιούνται περισσότερο οι άντρες. Ε, αυτοί οι τομεί όμω δίνουν και καλύτερη επαγγελματική εξασφάλιση. Οι περισσότερε γυναίκε δουλεύουν σε κοινωνικού τομεί που επηρεάζουν λιγά, λίγο, λιγότερο ε, τα, τα πράγματα και έχουν χαμηλότερου μισθού. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, να λάβουμε υπόψη μα το γεγονό ότι επειδή έχουν τη θέση που έχουν στην ε, στην οικογένεια οι γυναίκες για να έχουν οικονομική ανεξαρτησία να κάνουν σωστές σπουδές κτλ. Ε, το σημαντικό είναι να μην σταματήσει την ε, καριέρα της μια γυναίκα λόγω της α, οικογενειακής ζωή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ευέλικτη και συνεχή εκπαίδευση. Με αυτή την ε, έκθεση θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα και τα κοινωνικά εμπόδια που φράσουν τον δρόμο των γυναικών. Θέλουμε να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, ούτω ώστε να είναι στο επίπεδο των φιλοδοξιών των ε, κοριτσιών και να του δώσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην ισότητα των φίλων και στην ε, εκπαίδευση ε, και την σεξουαλική υγεία. Και θα πρέπει να σταματήσουν οι σεξιστικέ συμπεριφορέ στα σχολεία μα, που υπάρχουν και στην κοινωνία μετά. Ένα σχολείο, μία, ένα κορίτσι και, ένα, μια πένα μπορεί να αλλάξουν τη ζωή μιας γυναίκας. Υπόθηκε στην συνέλευση του ΟΗΕ για τους νέους ε, από ένα κορίτσι. Είναι σημαντικό αυτό να γίνει πραγματικότητα για όλα τα κορίτσια της Ευρώπης και του κόσμου. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σεντρό και ο κύριος Γουόρτ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εισαγωγή αυτή και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα δεν είναι πρόβλημα. Σήμερα τα κορίτσια, οι γυναίκες ολοκληρώνουν τις σπουδές τους ολοκληρώνουν την ανώτερη και την ανώτατη εκπαίδευση και μάλιστα σε μεγαλύτερα ποσοστά από ότι τα αγόρια. Το 60% των φοιτητών είναι γυναίκες. Άρα υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου και μάλιστα περισσότερες από ότι οι άνδρες ίδιας ηλικίας. Ποια είναι όμως η διαφορά. Αυτή εντοπίστε σε ένα διαφορετικό επίπεδο στα ανώτατα κλιμάκια, στα διευθυντικά στελέχη σχολείων και επιχειρήσεων. Εκεί είναι αντίστροφα τα ποσοστά. Και δεν σημαίνει αυτό ότι δεν ενδιαφέρουν οι θέσεις ευθύνη στις γυναίκες, αλλά υπάρχουν κάποια στάδια της επαγγελματική σταδιοδρομίας που μπορεί να διαφέρουν ε, οι φιλοδοξίες τους ε, ή οι σκοποί τους. Παραδείγματος χάρη αποκτούν παιδιά Οπότε ανακόπτεται η επαγγελματική τους εξέλιξη για κάποιο καιρό. Και στρέφονται σε άλλες δραστηριότητες διαφορετικές. Όταν μιλάμε λοιπόν για τη στήριξη των κοριτσιών και των γυναικών, φυσικά και μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την εκπαίδευση τους όμως, αν θέλουμε, να βελτιώσουμε και τη θέση που έχουν στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια συμφιλίωση και καλύτερη εναρμόνιση του οικογενειακού και του επαγγελματικού τους βίου. Σε ό,τι αφορά τώρα τα στερεότυπα των φίλων. Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα σχολεία, η πλειοψηφία είναι δασκάλες ε, μιλάω για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημοτικά και γυμνάσια. Οι περισσότερες ε, εκπαιδευτικοί είναι γυναίκες και μάλιστα αμείβονται χαμηλότερα. Είναι οι εκπαιδευτικοί που θα αναθρέψουν τη μελλοντική, τις μελλοντικές γενιές. πρέπει να δείξουν αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνουν άλλωστε την ε, ανατροφή και τη διάπλαση παιδιών, αγοριών και κοριτσιών. Υπάρχουν γυναίκες ε, που κάνουν αυτή τη δουλειά, άντρες δεν θα ήθελαν να την κάνουν επειδή είναι πιο χαμηλή αμοιβή όμως. Αυτά είχα να πω. Παρακαλώ ένα λεπτό οι επόμενοι ομιλητέ, γιατί αλλιώ είναι αδύνατο να ολοκληρώσουμε την ε, ημερήσια διάταξη. Τζούλη. Ευχαριστώ. Ως, μέλη, ως μέλος των Επιτροπών και Πολιτισμού και Γυναικών και υπερασπιστής των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών χαίρομαι που αναλαμβάνει πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Μαραγκάλ. Πρέπει πράγματι να σταματήσει αυτό το κενό στην εκπαίδευση. Στο επίπεδο του Πανεπιστημίου δίνεται η δυνατότητα στις γυναίκες να συμμετάσχουν καλύτερα στην κοινωνία και έτσι μειώνεται ο κοινωνικός αποκλεισμός με ό,τι αυτό σημαίνει για την υγεία, την ποιότητα ζωής και για τα κορίτσια και για τις γυναίκες. Η έννοια της ενδυνάμωσης των κοριτσιών έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης όπως η αυτοεκτίμηση είναι ε, κυριότερα χαρακτηριστικά των αγοριών. Τα αγόρια θεωρούν πως ε, τα ίδια είναι υπεύθυνα για την επιτυχία τους, ενώ για την αποτυχία ευθύνεται η κακοτυχία. Ε, σε αντίθεση με τις κοπέλες, οι οποίες υποτιμούν τις δυνατότητες τους. Και βεβαίως υπάρχουν και θέματα διαρθρωτικά και αυτά τα οποία αφορούν ε, την κοινωνία και το πώς βλέπει τα φύλλα. Οπότε συνολικά υπάρχει μια δομή η οποία ευνοεί τα αγόρια και μέχρι να ανατραπεί δεν θα υπάρξει πραγματική ισότητα. Οπότε θεωρώ πως η γνωμοδότηση του κυρίου Μαργκάλ είναι προς σωστή κατεύθυνση και εγώ προσωπικά συμφωνώ με το όραμα αυτό. Καλωσορίζω ιδιαίτερα την έμφαση που δίνεται στην ανάγκη να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα, το ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν ε, οι κοπέλες να ακολουθήσουν τις θετικές επιστήμες καθώς επίσης και η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην εκπαίδευση ενηλίκων, η εκπαίδευση των δασκάλων, τα σωστά πρότυπα που πρέπει να υπάρχουν γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά τα πρότυπα υπάρχουν ε, μόνο στερεότυπα και μετά ακολουθούν διάφορα άλλα προσβία. και τέλος ως και ο εγώ θα ήθελα να τονίσω το εξή η συμμετοχή των κοριτσιών στη δημοκρατική διακυβέρνηση των σχολείων πρέπει να υπάρξει ένα σωστό περιβάλλον για όλους τους μαθητές ε, και στο περιεχόμενο της διδακτέας ύλης, αλλά τα κορίτσια ιδιαίτερα πρέπει να μάθουν για τα δικαιώματά τους και να διδαχτούν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ζητήματα επίσης ε, σεξουαλικής αγωγής ε, και υγιεινής, ε, αλλά πρέπει να μάθουν ταυτόχρονα μαζί αγόρια και κορίτσια το τι είναι μια υγιή σχέση, ο σεβασμός, η αμοιβαιότητα και έχω και άλλα, έχω και άλλα. Έχουμε άλλους τρεις ομιλητές, είναι αδύνατο ε, να του ακούσουμε όλους, ειδικά αν όλοι μιλάνε τόσο. Ζητώ συγγνώμη, Τζούλη. Δεν γίνεται αλλιώ. Κύριος Κανεσδέσκι. Αντικαθιστά ένα σκιώδη Γιατί Ένα λεπτό όμως, σας παρακαλώ το πολύ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω κι εγώ πως ε, και θα διαβάσω την ε, δήλωση της κυρίας ε, Κασνιέσκα η οποία επίσης είναι μέλος της Επιτροπής Γυναικών άντρες και γυναίκες έχουν ίδια δικαιώματα το φύλλο δεν είναι μια τεχνητή κοινωνική επινόηση δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το ότι υπάρχουν διαφορετικά φύλλα η Κομισιόν με το να προωθεί αυτή την πολιτική, προωθεί μια πολιτική η οποία γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη. Από την εποχή του κομμουνισμού είχαμε να δει, είχαμε να δούμε στην Πολωνία τέτοια ιδεολογική πίεση. Το ότι δηλαδή το φύλλο έχει κοινωνική διάσταση είναι μία μέθοδος ε, προπαγάνδας ε, ε, στα νέα παιδιά και έτσι προωθείται ένα κοινωνικό μοντέλο. Γνωρίζουμε τώρα πως ε, περισσότερες γυναίκες αποφυτούν ε, από τα πανεπιστήμια και εκπαιδεύονται. Η πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας δίνει στις γυναίκες την δυνατότητα να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία το φύλλο δεν αποτελεί εμπόδιο στην εκπαίδευση. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι να κάνει διαθέσιμη την γνώση και τις δεξιότητες και έτσι καταπολεμάται η ανεργία και μπορεί κανείς βεβαίως να έχει μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Οι γυναίκες δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, χρειάζονται κάποια στήριξη για να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη γιατί έχουν πολλούς ρόλους να παίξουν στη ζωή. Σας ευχαριστώ για τη συντομία σας. Ευχαριστώ και την Κομισιόν. Ε, πρέπει 5 και 25 να αφήσουμε την αίθουσα και έχουμε ακόμα δύο γνωμοδοτήσεις. Ζητώ συγγνώμη ε, και από τον εκπρόσωπο των, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα του δώσω το λόγο σε μια άλλη ευκαιρία. Και τώρα, Κύριε Μαραγκάλ, μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη γνωμοδότηση, αν γίνεται. Θέλετε να πείτε κάτι έτσι, δύο τελευταία λόγια. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα έχουμε συζήτηση, θα ξανακάνουμε συζήτηση για αυτό το θέμα, από ό,τι βλέπω. Συμμεριζόμαστε πολλά θέματα. Βεβαίως υπάρχουν και στοιχεία θέματα στα οποία διαφοροποιούμαστε. Το ρόλο της κοινωνίας, του εκπαιδευτικού συστήματος κτλ. Ακούσαμε διάφορα από τους ομιλητές. Νομίζω ότι οι τροπολογίε θα μα δώσουν να εμπλουτίσουμε την έκθεση και να κάνουμε μια πιο ενδελεχή συζήτηση. Μιλάμε για ελευθερία. Μιλάμε για χειραφέτηση των γυναικών. Μιλάμε για πλήρη ανάπτυξη όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών τη Ευρώπη και του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης. Πρέπει να αλλάξουμε τα αντρικά στερεότυπα που επικρατούν. Όχι να τροποποιήσουμε τα θηλυκά στερεότυπα, αλλά και οι μεν και οι δε και οι άντρε και οι γυναίκε να καταλάβουν ότι μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο ελευθερία και ευθυνών ω υπεύθυνοι πολίτε. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε λύσει το θέμα τη ε, πρόσβαση στην εκπαίδευση. Όλοι τώρα έχουμε αυτό το δικαίωμα αλλά πρέπει να κατακτήσουμε ε, και το θέμα της κινητικότητας. Ε, επίσης, ε, η μετανάστευση προκαλεί νέες δυσκολίες στον τομέα αυτό. Να, πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε σωστά πρότυπα για τα κορίτσια, για το δημοτικό, για το γυμνάσιο, να τα προωθούμε στις επιστήμες. Να μην τους λέμε θα γίνετε γιατροί μόνο οι δασκάλες. Και επίσης, το το να είσαι γυναίκα θα πρέπει να το συνδέουμε με την έννοια της κοινωνικής ευθύνης. Επίσης θα πρέπει να ανακαλύψουμε το ταλέντο που μπορεί να έχουν ε, γυναίκες για επιστημονικούς κλάδους, ε, μηχανικούς κλάδους κτλ. Πρέπει να έχουμε θετικά γυναικεία πρότυπα. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κυρία Μαραγκάλ. Είναι τόσο ωραία αυτά που λέτε για τις γυναίκες. Πραγματικά πονάω, πονάει η ψυχή μου που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να το κάνω. Ε, χαίρομαι για αυτή την πρωτοβουλία που, προκαλεί, που προωθεί η ε, Επιτροπή Γυναικών, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι έχουμε αφήσει το θέμα σε τέλεια χέρια, στα καλύτερα χέρια. Οι τροπολογίες. Μέχρι τις 30 Μαρτίου 12 η ώρα. Πάμε στο επόμενο θέμα, πάρα αυτά, στην έκθεση του σχεδίου γνωμοδότηση για τη δημιουργία μια ανταγωνιστική αγορά εργασία που και τον πρώτο, ε, 21ο αιώνα αντιστοίχηση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τι ευκαιρίε. Ε, θα ψηφίσουμε στις 5 Μαΐου, 12.30, συγγνώμη, πάλι 30 Μαρτίου, ε, έχουμε προθεσμία 12, 12 η ώρα για την υποβολή των ε, τροπολογιών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, μια ανταγωνιστική αγορά εργασία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 21ο αιώνα είναι κορυφαία προτεραιότητα της Ένωσης, αλλά ο μόνος ενωση αλλα ο μονος τροπος να επιτευχθεί είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ δεξιοτήτων και προσόντων. Και έτσι θα ε, μειωθεί η ανεργία των ε, νέων, θα ανακάμψει ε, γρήγορα η Ευρώπη και θα έχουμε βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των εξής σημείων. Θα συνεχιστεί η τάση, οι θέσει εργασία να γίνονται όλο και πιο απαιτητικέ γνώσει. Το 2020 η πλειοψηφία των θέσεων εργασία που δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαιτεί ε, μέσα ή υψηλά προσόντα. Ο κόσμος που ε, δεν θα τα έχει θα δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να βρει μια δουλειά. Οπότε το ζήτημα αυτών των δεξιοτήτων πρέπει να είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμιστούν οι δεξιότητες με τις ανάγκες της ε, αγοράς εργασίας επενδύοντας σε ψηφιακές δεξιότητες, σε γλωσσικές ικανότητες ε, και βεβαίως ε, το θέμα της Ευρώπης ε, αλλά και της προσωπικής εξέλιξης είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ανταποκριθούμε στις δουλειές που θα δημιουργηθούν το μέλλον, στο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα της ε, άτυπης και ανεπίσημης εκπαίδευσης ε, επίσης πρέπει να τονιστεί η δυνατότητα να αποκτήσει κανείς πρακτικές δεξιότητες ε, έχει μεγάλη σημασία εγκάρσιες δεξιότητες επίσης που έχουν μεγάλο πεδίο εφαρμογής η εσωτερική κινητικότητα επίσης πάρα πολύ σημαντική η βελτίωση των δυνατοτήτων κινητικότητας καθώς και η βελτίωση των στρατηγικών ε, πρόσληψης ε, και εκπαίδευσης. Τέλος, η έκθεση επίσης ε, τονίζει την σημασία της αναγνώρισης ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων σε διεθνές επίπεδο καθώς και ε, της εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για το να είναι, είναι σε θέση να βρουν μια θέση εργασία στην ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ. Δύο άτομα θέλουν τον λόγο. Η κυρία Τρούπελ που είναι σκιώδη συγγήτρια και η κυρία Τζούλι Γουόρντ αντί για τον κύριο Μίτσι. Very briefly, um... Ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα. Στην τελευταία περίοδο αλλά και πιο πριν ακόμη είχαμε μια έκθεση για τις βασικές δεξιότητες για τη διαβίου μάθηση και πάνω σε αυτά τα απορίσματα πρέπει να οικοδομήσουμε. Ήταν σαφές ε, ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες, άρα ένα είδος follow-up πρέπει να κάνουμε, όχι να επανεφεύρουμε από την αρχή τον τροχό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Τζούλη σύντομα. Εκπροσωπώ τη συνάδελφο Μαρλίν Μίτσι τον συνάδελφο μάλλον. Η έκθεση του κ. Κιουτσούκ, ε, η γνωμοδότησή του είναι ισορροπημένη, κάνει πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, να επενδύσουμε δηλαδή ε, Στι εκπαιδευτικέ δεξιότητες, να τονίσουμε την άτυπη ε, εκπαίδευση, το Erasmus Plus και να συμπληρώσουμε τα μέτρα ε, με στόχο την αντιμετώπιση της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου και της ανεργίας των νέων. Δεξιότητες λοιπόν, θέσεις εργασίας. Πολλές φορές θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε σε νέες δεξιότητες, στις νέες τεχνολογίες Θέλει έρθω λοιπόν να πούμε ότι η έλλειψη δεξιοτήτων, το έλλειμμα δεξιοτήτων μπορεί να μην αυξάνει άμεσα ε, την ανεργία. Αυτό το πράττει η οικονομική κατάσταση, η οικονομική κρίση που οδηγεί σε υποαπασχόληση ανεργία. Δεν υπάρχει όμως καλή αντιστοίχηση δεξιοτήτων. Αυτό έχει να κάνει και με άτομα που έχουν πάρα πολύ μεγάλα προσόντα, αλλά δουλεύουν ε, σε πιο χαμηλές θέσεις, με χαμηλότερη ειδίκευση. Δεν μπορούμε λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με την αντιστοίχηση των δεξιοτήτων και των προσών. Σίγουρα όμως πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες αυτές. Να προσαρμοστούμε στις μελλοντικές τάσεις της αγοράς, γιατί οι νεότερες γενιές μπορεί να πληρώσουν τα δικά μας λάθη. Θέλουμε και βραχυπρόθεσμα μέτρα και μακροπρόθεσμες στρατηγικές για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι νέοι τις δεξιότητες για το μέλλον που θα τους βοηθήσουν στον επαγγελματικό τους ε, βίο. Θέλουμε μια ολιστική προσέγγιση για τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, ε, να μειωθεί το πρόβλημα της αντιστοίχησης των δεξιοτήτων με τη ζήτηση, για να μπορέσουν να ευημερίσουν νέοι στην... Έχει πολλά, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, είναι πάρα πολλές οι υποδείξεις, πολύ καλές. δεν το δίνετε το χαρτί κατευθείαν στον εισηγητή. Ναι, είναι δολογική η προσέγγιση πάντως και είναι, είναι σημαντική. Ναι, είναι σημαντικό, αλλά δώστε το χαρτάκι στον εισηγητή, καλύτερα. Θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Είναι πολύ πολύ ζητώ συγγνώμη από την Κομισιόν. Αλλά μέσα σε 10 λεπτά που μα μένουν πρέπει να ολοκληρώσουμε ε, και το επόμενο θέμα και να μεταβούμε στην άλλη αίθουσα που πρέπει να είμαστε στις 5.30 όπου έχουμε την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ah, ok. Ehm, maybe that we are, allora, I imagine that, eh, caro collega Morgano. Κύριε Μοργάνο, μήπως θα μπορούσαμε να αναβάλουμε τη δική σας έκθεση. Έχουμε τη δυνατότητα του Μαΐου. Μπορούμε, βεβαίω. Και μπορούμε να το συζητήσουμε με την ησυχία μας. Επομένως, η Κομισιόν, αν θέλει κάτι, μπορεί να το πει. Αλλιώς μπορούμε να εγκαταλείψουμε την αίθουσα τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μαρία Κιάρα Ριουντίνο, λέγομαι. Δουλεύω στην Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, ε, Δεξιότητε και Προσόντα, στο τμήμα Δεξιότητε και Προσόντα. Θα είμαι συντομότατη. Καλωσορίζουμε το σχέδιο γνωμοδότηση. Πιστεύουμε ότι τα σημεία που αναφέρονται στο σχέδιο έκθεση είναι ουσιαστικά εντός θέματος απόλυτα. Περιμένουμε τη συνεργασία με την Επιτροπή σας και με την Επιτροπή Απασχόλησης. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την κατανόηση και την Κομισιόν. Νομίζω είναι μια σημαντική έκθεση αυτή, γιατί αποτελεί συνέχεια ε, των εκθέσεων που έχουμε ετοιμάσει για την ενίσχυση των δεξιοτήτων. Λοιπόν, να δύο πράγματα. Τώρα θα πάμε στην αίθουσα. 2 Γιάν 2 για τη συνάντηση με την ε, Επιτροπή ΑΦΕΤ. Αύριο το πρωί στις 9 και κάτι θα ξεκινήσουμε τις ε, ψηφοφορίες. Επομένως, να έχετε την κάρτα ψηφοφορίες σας μαζί, έτσι. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην αίθουσα 2Q2 και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας. Και ευχαριστώ και τους ε, εισηγητές εννοείται.